Possiamo iniziare? Να ξεκινήσουμε. Θα περάσουμε στην ψηφοφορία διανατάσσεως χειρός μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν κριθεί απαραίτητο, θα χρησιμοποιήσουμε την ε, ηλεκτρονική επαλήθευση και θα ψηφίσετε με τις κάρτες σας. Να σας πω ότι όλες οι ομάδες έχουν συμφωνήσει και για τις τελικές ψηφοφορίες, επομένως θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε χάρη στη συμφωνία αυτή, ελπίζω ακόμα πιο γρήγορα. Έτοιμοι λοιπόν. Άλμπερτ, μήπως θέλεις να πεις κάτι πριν ψηφίσουμε? No, bene, avanti. Ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν. Μπορούμε να προχωρήσουμε. Tutti pronti? Allora, iniziamo... Έτοιμοι λοιπόν. Ξεκινάμε την ψηφοφορία. Κοινή αγροτική πολιτική για το 2020. Διανατάσεως χειρός. Υπέρ της συμβιβαστικής τροπολογίας παριθμών 1. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα, διανατάσσεως χειρός πάντα, τη συμβιβαστική τροπολογία 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 3. Μισό λεπτό, συγγνώμη. Ψηφίζουμε την τροπολογία 231 με ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται ψηφοφορία. Ηλεκτρονική ψήφος. It doesn't work. Apri. Apri voto. Eh. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. Έχουμε δύο ψήφους επιπλέον, μία από το ΕΛΚ και μία από τους σοσιαλιστές. Δύο επιπλέον ψηφίζουν. Παρακαλώ. Ξαναψηφίζουμε λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 231. Πε... Πέρασε ψηφοφορία. ψηφοφορία. και πάλι υπάρχει μία επιπλέον ψήφος του ΕΛΚ. Εγκρίνεται παρόλα αυτά, σας παρακαλώ ελέγξτε όμως ποιοι ψηφίζουν. Περνάμε τώρα στη συμβιβαστική τροπολογία 3. Δυνατά χειρό. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. με ηλεκτρονική επαλήθευση την 267. Άρχεται η ψηφοφορία 267. Ψήφισαν όλοι για τη 267 πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 272. Ψήφισαν όλοι. Πέραση της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Διανατέσεις ο χειρός τώρα συμβιβαστική τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 6. υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχ... Κατά αποχές εγκρίνεται. «381 ηλεκτρονικός». «381». Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τη συμβιβαστική τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Με ηλεκτρονική επαλήθευση θα ψηφίσουμε τώρα την 497. 497. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 17β με ηλεκτρονική ψήφο. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Για τη συμβιβαστική τροπολογία 17β. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε τώρα, διανατάσσεως χειρός, συμβιβαστική τροπολογία 18, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 19, διανατάσσεως χειρός πάντα, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Unblock τώρα ψηφίζουμε τις... Unblock λοιπόν ψηφίζουμε τις 20 έως 23 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τώρα περνάμε με ηλεκτρονική ψήφο την 643. Άρχεται η ψηφοφορία για την 643. 643 ψήφισαν όλοι. Πέραση ψηφοφορία. Απροβάτο. Εγκρίνεται. Περατζάτα τη Προχωράμε. Συμβαστική τροπολογία 24. Υπέρ. Και κόντρο. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 25. Διανατάσσεως χειρός και πάλι. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε σε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την 478 Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. 478 απορρίπτεται. Πάμε τώρα στην 500. Άρχεται η ψηφοφορία για την 500. Votato tutti, chiuso 500. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συνεχίζουμε. 692. Άρχεται η ψηφοφορία για την 692. Πέρασε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα την 752. Άρχεται η ψηφοφορία για την 752. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 756. Άρχεται η ψηφοφορία για την 756. Ψήφισαν όλοι, πέρασε της ψηφοφορίας. Η 756 απορρίπτεται. 757. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Απορρίπτεται η 757. 759. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 758. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 754. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 755. Άρχεται η ψηφοφορία για την 755. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Και τέλος η 760. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Διανατάσσεως χειρός και πάλι. Συμβιβαστική τροπολογία 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 27. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 784 με ηλεκτρονική επαλήθευση άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η 784. Διανατάσσεω χειρός και πάλι. Συμβιβαστική τροπολογία 28. Άρχεται η ψηφοφορία. Υπέρ, συγγνώμη κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την 853 ηλεκτρονικός. Άρχεται η ψηφοφορία για την 853. Κατά, συγγνώμη, ψήφισαν όλοι για την 853 πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Per votazione Ηλεκτρονικά. Ψηφίσουμε την 892. Άρχεται η ψηφοφορία για την 892. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 894. Άρχεται η ψηφοφορία για την 894. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συνεχίζουμε. Συμβιβαστική τροπολογία 38. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 43. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 44. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την παράγραφο 45 ηλεκτρονικός ενοποιημένη τροπολογία που προτείνεται από τον εισηγητή άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε τη 45. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέραση τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε τώρα ηλεκτρονικός ψηφίζουμε τη 1022. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 1022. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονικά την 1023. 1023, προσοχή, 1023 πατράω. Άρχεται η ψηφοφορία. Chiusa la votazione. Πέρασε τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1025. 1025 με ηλικιωτική ψηφοφορία. 1025. Πέραση τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Παράγραφος 46. Ενοποιημένες τροπολογίες που προτείνει ο εισηγητής. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και τέλος, και πάλι ηλεκτρονικό στη 1035. 1035, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και τώρα. Συνεχίζουμε δυνατό ω χειρός. Συμβαστική τροπολογία 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονικά τώρα. 1052. 1052. Εράντς και άλλοι. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε τη ψηφοφορία, εγκρίνεται. 1043. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 1043. Πέρασε τη ψηφοφορία. εγκρίνεται. Διανατάσσεω χειρό και πάλι. Συμβιβαστική τροπολογία 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 48. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 49. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε. Συμβαστική τροπολογία 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. με ηλεκτρονική επαλήθευση τώρα άρχεται η ψηφοφορία για τη 1094. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 1094. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 51 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 52 υπέρ κατά κατά εγκρίνεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία τώρα για τη 1029, 1129 άρχιτη ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται. Διανατάσεως η συμβαστική 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 57 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβασ... Μάλλον ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρθρη ψηφοφορία για την τροπολογία 1227. Άρθρη ψηφοφορία. Ψηφιστόλη. Πέρας εγκρίνεται. Διανατάσσος ισχυρός τη συμβαστική τροπολογία 59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία στη συνέχεια για την ε, τροπολογία 1235. 1249 με συγχωρείτε. Πέρας. Ζητώ συγγνώμη, άρχεται η ψηφοφορία για τη 1235, διορθώνει ο πρόεδρος, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τη 1235, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. «1238». Ναι, ναι. Άρχεται ψηφοφορία για τη 1238. Δαντάμ, Παπαστάκομς, πέρας. Εγκρίνεται. Άρχεται ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 1240 Ντόρφμαν. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη 1240. Πέρας. Εγκρίνεται. «1241». Άρτη ψηφοφορία για τη 1241. Πέρας. Εγκρίνεται. Διανατάσσου χειρό τώρα, συμβαστική τροπολογία 60 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τρο... πρόεδρος. Συμβαστική τροπολογία α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία Bα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία E υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία F υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία G υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία GA υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία GB υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία H υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία I υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία IA υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 101, άρτη ψηφοφορία για την 101, έραντς και άλλοι. Ψηφίστε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε διανατάσσος χειρός, συμβαστική τροπολογία και υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία LA υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία LB υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία M υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία ο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία π υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία PA ε, υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία PB υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία PC υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Θα ψηφίσουμε τώρα on bloc τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι πολιτικές ομάδες. Θα ψηφίσουμε όλα τα citations μαζί, όλες οι τολικές αναφορές δηλαδή, υπέρ on block ψηφίζουμε, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Συνεχίζουμε τώρα. Πρέπει να ψηφίσουμε τις γνωμοδοτήσεις των άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών Διανατάσεις ισχυρό πάντα. Δεβε αλφα υπέρ. Σε συγγνώμη, δεβε έξι με συγχωρείτε, ΔΕΒΕ 6 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. ΔΕΒΕ 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. NV20 υπέρ, Κατά. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την MV20. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. NV27. Συνεχίζουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Θα προχωρήσουμε πια πιο γρήγορα. NV27 λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. NV28, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάντα με ηλεκτρονική ψηφοφορία ψηφίζουμε την NV29, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. NV31. Άρτη ψοφορία. Πέρας. εγκρινεται nv MV35. Άρχεται ψοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. MV40. Όχι, καταπίπτει αυτή. Ψηφίζουμε την Ήτρε 6, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ήτρε 9, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ήτρε 15. Εγκρίνεται η Ήτρε 9. 29 προς 15. Ήτρε 15 τώρα. Άρτε ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ήτρε 16. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ήτρε 17. Άρχεται η ψηφοφορία για την Ήτρε 17. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην Regi 5. Άρχεται η ψηφοφορία για τη Regi 5. Πέρας. Γκρίνεται. Regi 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίστε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Ρέτζι 17. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τελική τώρα ψηφοφορία για το σύνολο της έκθεσης όπως τροποποιήθηκε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε η ψηφοφορία, πέρας. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας. Με τέσσερις αποχές και μία μόνο ψήφο κατά, 40 υπέρ, συγχαρητήρια κύριε Ντές. Rimanete qui che Στις θέσεις σας για να ψηφίσουμε πολύ γρήγορα και τι υπόλοιπε εκθέσει. Να δώσουμε όμω πρώτα το λόγο στον Άλμπερτ Τέσ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, μετά από αυτήν την ψηφοφορία θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους, όλους που στηρίξατε αυτές τις συμβιβαστικές τροπολογίες Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους ε, συντονιστές, τους κοιόδες εισηγητές, αλλά βεβαίως και όλους τους συναδέλφους οι οποίοι έχουν συνεισφέρει στην προετοιμασία και στην τροποποίηση αυτής της έκθεσης με τις προτάσεις σας, ιδιαίτερα στην δική μου ομάδα, όπου πολύ συζητήσαμε. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα Νομίζω ότι στέλνουμε ένα πολύ συγκεκριμένο μήνυμα στον Επίτροπο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίρνει θέσεις συγκεκριμένες ε, για το ποια θα είναι η κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε κυρίως μετά το 2013 και ότι η Επιτροπή επίσης θα πρέπει να δει ότι με μεγάλη πλειοψηφία στηρίχτηκε η έκθεση αυτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μπορούμε να συνεχίσουμε λοιπόν τις εργασίες μας τώρα. Σημείο 13 στην ημερήσια διάταξη, τροποποίηση του κανονισμού 834-2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων. Μάρτιν Χάουσλινγκ ο εισηγητής. Ξεκινάμε λοιπόν η πρόταση έχει περιοριστεί μόνο στι απαραίτητες τροποποίησεις για την ευθυγράμμιση του κανονισμού. Ο εισηγητή υποστηρίζει με σθένο την πρόταση τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρουσιάστηκαν 23 τροπολογίες στο σύνολά 13 από τον εισηγητή και εγκρίνουν κυρίως ε, άρθρα που αφορούν ε, το κοινό πνεύμα μεταξύ των θεσμικών εργάνων και την κοινή συμφωνία για τις εκτελεστικές πράξεις και τις πράξεις κατεξουσιοδότησης. Υπάρχει κατάλογος ψηφοφοριών. Αν ο Μάρτιν δεν θέλει το λόγο μπορούμε να ξεκινήσουμε μέσα στη ψηφοφορία. Ο Μάρτιν δεν θέλει το λόγο. Ωραία. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 16. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 16. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε της ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 17. Πέρασε της για την τροπολογία 17. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία για την 4. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της Εγκρίνεται. Άρχεται η ψηφοφορία για την 5. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της Εγκρίνεται. 18. 6, συγγνώμη, τροπολογία 6, άρχεται η ψηφοφορία. Απροβάτο. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Άρχεται η ψηφοφορία για την 7. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε τις ψηφοφορία για την 7. Εγκρίνεται. Το 19. Τροπολογία 19. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε τις ψηφοφορίες για τη 19. Απορρίπτεται. Έχουμε δύο επιπλέον που ψηφίζουν για το ΕΛΚ. Σας παρακαλώ προσέξτε λίγο τις ψήφους σας. Δύο επιπλέον ψήφους για το ΕΛΚ. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 21. Τροπολογία 21. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Unblock. Άρχεται η ψηφοφορία. Η 9, 10, η 11 και κάποιες από τις αιτιολογικές σκέψει πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Το μπλοκ τροπολογία 20. Άρχεται η ψηφοφορία για την 20. Chiusa la votazione sul 20. Πέρας της ψηφοφορίας για το 20. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. εγκρίνεται. Και τέλος, 15. Ψηφοφορία για τη 15. Ψήφισαν όλοι. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ψηφίσουμε τώρα την νομοθετική πρόταση ως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία για την νομοθετική πρόταση. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το νομοθετικό ψήφισμα. Ψήφισαν όλοι. Πέρας εγκρίνεται και τέλος ψηφίζουμε την εντολή για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Άρχεται η ψηφοφορία για τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια Μάρτιν. Προχωράμε παρακάτω. Σημείο 14. Ορισμένοι συνάδελφοι πρέπει να ψηφίσουν στην ΣΟΥΡΕ. Επομένως, ή δυνατόν να αντιστρέψουμε λίγο τη σειρά με την σύμφωνη λοιπόν γνώμη σας να ψηφίσουμε ευθύ αμέσω ε, την έκθεση Λαβία, τη σχέδιο γνωμοδότησης Λαβία. Επομένω περνάμε στο σημείο 16. Συμφωνείτε. On block μπορούμε να ψηφίσουμε όλες τις α, τροπολογίες της έκθεσης Λαβία, τροποποίηση του κανονισμού 1290-2005 του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία on block, ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται συγχαρητήρια στον κύριο Λαβία. Πηγαίνετε να ψηφίσετε τώρα στη ΣΟΥΡ και προωθήστε εκεί, περασπίστε τη στάση της δικής μας Επιτροπής. Πρέπει να κάνουμε και άλλες δύο ψηφοφορίες όμως. Ακολουθώντας τη διαδικασία ψηφίζουμε την νομοθετική πρόταση όπως τροποποιήθηκε. Είναι η τελική ψηφοφορία πρέπει να γίνει σε σχέση με την έκθεση αυτή. Ψηφίσατε όλοι για την νομοθετική πρόταση. Πολύ ωραία πέρας και εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το, την, ε, το ψήφισμα, το νομοθετικό ψήφισμα. Άρχεται η ψηφοφορία για το νομοθετικό ψήφισμα. Εγκρίνεται. Και τέλος ψηφίζουμε την απόφαση για την ένταξη πραγματεύσεων με το Συμβούλιο. Ψηφίσατε όλοι. Πολύ ωραία. Έχουμε καλύψει έτσι και τις τυπικές διαδικασίες. Σας ευχαριστώ και επιστρέφουμε στο σημείο 14 τροποποίηση του κανονισμού του Συμβουλίου 485 του 2008 περί των ελέγχων εκ μέρους των κρατών μελών των πράξεων που αποτελούν μέρος του συστήματος χρηματοδοτήσεως από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγύσεων. Η συγητής είναι ο Λουίς Μάνουελ Κάπουλα Σάντος. Αν συμφωνεί ο εισηγητής μπορούμε να ψηφίσουμε on block. Συμφωνεί ο εισηγητής, ψηφίζουμε on block. Άρχεται η ψηφοφορία για την έκθεση Κάπουλας Σάντος. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την νομοθετική πρόταση όπως τροποποιήθηκε. Ψηφίσατε όλοι. Ψηφίζουμε τώρα το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος άρτη ψηφοφορία. Εγκρίνεται και τέλος ψηφίζουμε για την απόφαση έναρξης διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο. Πέρας. Εγκρίνεται. Πολύ ωραία συγχαρητήρια στον Λουίς. Σημείο 15 τροποποίηση του κανονισμού 378 του 2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες για την εφαρμογή της προαιρετικής διαφοροποίησης των άμεσων ενισχύσεων στα πλαίσια της κοινή γεωργικής πολιτικής. Η συγγήτρια κυρία Μπρίτα Ρέιμερς. Ρίτα, θέλεις το λόγο? Όχι. Συμφωνείς να ψηφίσουμε on block τις τροπολογίες. Ναι, πολύ ωραία. Άρχεται η ψηφοφορία on block για όλες τις τροπολογίες της κυρία Μπρίτα Ρέιμερ, της έκθεση κυρίας Μπρίτα Ρέιμερς. η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. η ψηφοφορία για την νομοθετική πρόταση ω τροποποιήθηκε. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος άρθρη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Και ψηφίζουμε για την απόφαση να ξεπραγματεύσουμε το Συμβούλιο. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται και το σημείο 15 συγχαρητήρια στην Μπρίτα Ρέιμερς. Αγαπητοί συνέδελφοι, ήταν πολύ σημαντική η σημερινή ημέρα. Είχαμε μια πολύ, καλή ακρόαση με τον κύριο Πρόντι και ψηφίσαμε και την έκθεση DES. Συγχαρητήρια σε όλους και θα τα πούμε στις 21 Ιουνίου στις 9 το πρωί.